χειρεύει και πρέπει να πληρωθεί. Ο κύριος Ρίχαρτ Ζούλικ έφυγε από την ομάδα ALDE και πήγε στην ομάδα ECR από τις 8 Οκτωβρίου 2014.